Παρακαλώ, καθίστε έτσι ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας όλο το χρόνο που θα μας αφιερώσει η Επίτροπος. Ξεκινάμε με την υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν διαφωνείτε, θεωρείτε ε, εγκεκριμένη ανακοινώση του Προέδρου, ε, γλωσσικό καθεστώς, διερμηνία πω και προς τα ελληνικά μεταξύ άλλων. Συστά συντονιστών, σύμφωνα με τον κανονισμό 205, Λαρόεντσο, εισηγητή Φοντάν από το ΙΕΝΕΦ, ε, εισηγητή για την έκθεση ε, απόφαση Συμβουλίου για την εφαρμογή ε, του συμφωνίας της ε, Europol για τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Βοσνίας Ζεγοβίνης και Ευρωπόλ. Συμφωνείτε με αυτή την ε, σύσταση των συντονιστών. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 3, το βασικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης. Ευχαριστώ πολύ που είστε παρόντες εδώ πολύ άριθμοι. Έχουμε μια σημαντική παρουσίαση της, ε, των απόψεων της Επιτροπής σχετικά με την απόφαση στην υπόθεση Maximilian Schrems ε, κατά του Επιτρόπου Προστασίας των Δεδομένων του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 6 Οκτωβρίου. Ε, καλωσορίζω την ε, κυρία Βέρα Γιουροβά, Επίτροπο Αρμόδια για τη Δικαιοσύνη στους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φίλων. Θα εστιάσουμε στην υπόθεση Schrems. Ε, θα κάνουμε και, δύο αναφορές, δύο ε, αναφορές, ανακοινώσεις για θέματα ε, ΛΟΑΔ και άλλα, αλλά στο τέλος αυτό. Στις 12 Οκτωβρίου η Νομική Επιτροπή ε, παρουσίασε την γνώμη της και τις εξελίξεις και είχαμε και μια πρώτη ενημέρωση από την Επιτροπή όμως σήμερα θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε την Επίτροπο για αυτή την απόφαση, να μας μιλήσει για αυτή την απόφαση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιουρόβα να μας κάνει την παρουσίασή της για την απόφαση αυτή του ε, Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά θα προχωρήσουμε σε λεπτομερή συζήτηση. Έχει το λόγο. you, like thank... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Λίμπε. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Ήθελα να ε, παρευρεθώ το νωρίτερο δυνατόν για να σας δώσω νέες πληροφορίες για τα βήματα τα οποία αναλαμβάνει η Κομισιόν σε σχέση με την απόφαση ΣΡΕΜΣ της 6ης Οκτωβρίου. Όπως ήδη είπα στην Ολομέλεια δύο εβδομάδες πριν, έχω δεσμευτεί να σας ενημερώσω, να σας ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα και θα ήθελα να με υποστηρίξετε σε αρκετά ζητήματα σε σχέση με την εργασία μας επί του θέματος αυτού. Θα επανέλθω αργότερα σε αυτό. Η συζήτηση στην Ολομέλεια έλαβε χώρα στις 14 Οκτωβρίου όπου αναφέρθηκα στις άμεσες προτεραιότητες της Επιτροπής μετά την απόφαση ΣΡΕΜΣ. Θα ήθελα να σας πω ποιες είναι αυτές οι προτεραιότητες, γιατί παραμένουν οι ίδιες. Να εγγυηθούμε στους πολίτες την προστασία προσωπικών δεδομένων όταν μεταφέρονται στο εξωτερικό, να υπάρχει διαφάνεια για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θα πρέπει να μεταφέρουν ε, πληροφορίες της ΕΠΑ και να εργαστούμε με τις εθνικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων για να μην υπάρχει κατακαιρματισμό στην εσωτερική αγορά της Ευρώπης. Επίσης, η Ευρώπη θα επιταχύνει τις συζητήσεις με ΕΠΑ για τις διατλαντικές ροές πληροφοριών. Θα συνεργαστώ μαζί σας ε, στα πλαίσια εταιρικότητας και διαφάνειας. Θα σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις και ελπίζω να ακούσω από εσάς πώς βλέπετε αυτή τη διαδικασία εν ώψη της επίσκεψής μου στη Ουάσιγκτον κατά τα μέσα Νοεμβρίου. Μετά τις 14 Οκτωβρίου στην Ολομέλεια η Επιτροπή συνεργάστηκε με τις Ευρωπαϊκές Αρχές, αρχές προστασίας δεδομένων, την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Δεδομένων, δυνάμει της ομάδας εργασίας άρθρου 29. Ο ρόλος αυτής, ε, αυτών των ανεξάρτητων αρχών τονίστηκε ιδιαίτερα στις 16 Οκτωβρίου η ομάδα εργασίας άρθρου 29 συνέταξε ένα κείμενο για τις συνέπειες της απόφασης. Αναφερθήκαμε στις συνεχόμενες ε, διαδικασίες μέσα στα πλαίσια των, ε, των διαδικαστών ασφαλούς λιμένα και μιλήσαμε για το ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα πρέπει να βρουν τρόπους μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ που να συνάδουν με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ως προς τις ροές προσωπικών δεδομένων, η ομάδα εργασίας έκρινε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και συμβατικές ρήτρες καθώς και επιχειρηματικές ε, ρήτρες έτσι ώστε να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των ε, μέσων. Η ομάδα εργασίας τόνισε ότι αν μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2016 δεν έχει εξευρεθεί λύση με τις αρχές των ΙΠΑ και με βάση την έκβαση της εκτίμησης των εναλλακτικών μέσων, η Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα επιβολής και θέσει σε ισχύ των νέων μέτρων. Θέλουμε ε, ε, μια νέα διατλαντική συμφωνία μέχρι τον Ιανουάριο του 2016. Θεωρούμε όμως ότι ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να ε, διακατέχεται από σαφήνεια. Όταν το συζητήσαμε με τους Άνσιπ και Έτιγκερ, τους, τους δύο επιτρόπους, στις 14 Οκτωβρίου, προσπαθήσαμε να έχουμε μία ενιαία ερμηνεία της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η Επιτροπή θα εκδώσει ε, μία ε, ανακοίνωση επεξηγηματικής φύσης ε, με βάση την απόφαση ΣΕΡΜΣ για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Αυτό δεν αντικαθιστά βεβαίως την εργασία των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Επιτροπή θα υποστηρίζει την εργασία τους έτσι ώστε να υπάρχει ενιαία προσέγγιση μέσα στα πλαίσια της ομάδας εργασίας του άρθρου 29. Θα ήθελα να πω επί της ουσίας σε σχέση με τις τρέχουσες διαδικασίες με τις ΕΠΑ το θέμα του ασφαλούς λιμένα ήταν μία από τις βασικές αρχές για τις μεταφορές δεδομένων από την Ευρώπη στις ΗΠΑ. Θα πρέπει όμως να μιλήσουμε για ένα νέο πλαίσιο δεδομένων με τις είπα για την ε, ροή δεδομένων διατλαντικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το διατλαντικό εμπόριο και βεβαίως και για τους πολίτες μας. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να τηρήσει τα δεδομένα της απόφασης ΣΡΕΜΣ. Αν και πριν από την απόφαση η Επιτροπή όρισε ζητήματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια των 13 συστάσεων του 13 για το Safe Harbor. Χρειαζόμαστε περισσότερες διασαφηνίσεις από τις αρχές των ΙΠΑ σε πολλά σημεία. Και φυσικά επιταχύναμε τη διαδικασία, δηλαδή ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τους ομολόγους των ΙΠΑ και έγιναν πολλές συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο. Μίλησα με τον Υπουργό Εμπορίου Σπρίκερ και τις επερχόμενες εβδομάδες θα γίνουν συζητήσεις σε τεχνικό επίπεδο και θα βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή πριν μεταβώ στην Ουάσιγκτον κατά τα μέσα Νοεμβρίου. Αυτές οι συζητήσεις δεν είναι καθόλου εύκολες, θέλω να με πιστέψετε, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει επιτελεστεί σημαντική πρόοδος. Θα πρέπει και θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι επιπτώσεις της απόφασης και πώς θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν αμφισβητεί τις εξουσίες της Επιτροπής να λάβει αποφάσεις επάρκειας. Διασαφηνίζει στοιχεία ως προς τις ε, ρυθμιστικές αρχές για να παρεύουν σε περίπτωση προσφυγών όπως εκείνη του κυρίου Σρέμς και παράλληλα να υπάρχει ένα επίπεδο προστασίας σε τρίτη χώρα κάτι το οποίο δεν είναι παρόμοιο αλλά εφάμιλο με το μέτρο ή τα μέτρα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο νεοεκλογής, νεοεκλεγής πρόεδρος του δικαστηρίου, κύριος Λέναρτς, είπε τα εξής ως προς την απόφαση Σρέμς. Η απόφαση δεν διακόπτει η κυρία Γιούροβα. Εξήγησε ότι το δικαστήριο δεν αποτιμά το σύστημα των ΙΠΑ καθώς και το σύστημα πληροφοριών του. Και τώρα έρχεται το παράθεμα. Κρίνουμε το την ενδοκινοτική νομοθεσία σε σχέση με τη μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες. Η απόφαση δεν σημαίνει ότι θα αναγνωρίσουμε το σύστημα, το νομικό σύστημα των ΙΠΑ. Όταν μιλάμε όμως για μεταφορά ε, δεδομένων, θα πρέπει να υπάρχουν ε, ρήτρε διασφάλισης που να είναι ισόνομες με αυτές της Ευρώπης. Αυτό αποζητώ και στη συζητήσεις μου με τις αρχές των ΙΠΑ. Το δικαστήριο τονίζει ότι η αυτοπιστοποίηση τύπου safe harbor είναι αποτελεσματική τη στιγμή που υπάρχει σωστή εποπτεία και ανείχνευση των προβλημάτων. Αυτό ήταν ένα σύστημα, ζήτημα μάλλον κλειδί που μας απασχόλησε με τους ομολόγους των είπα μετά από τις συστάσεις ε, του Νοεμβρίου του 2013 1-2 του για την διαφάνεια και για, τις, για την αποκατάσταση γιατί το εμπορικό επιμελητήριο παρέβλεψε ορισμένα στοιχεία, γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προσφυγές από, την, από το Ομοσπονδιακό Εμπορικό Επιμελητήριο. Έτσι θα υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να έχουμε να κάνουμε με ένα ενεργό σύστημα και με την ενίσχυση των κυρώσεων. Γι' αυτό θα θέλαμε οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων να είναι προενεργές και πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Εργαστήκαμε για τη βελτίωση των σημείων διεπαφής μεταξύ εθνικών αρχών και εμπορικού επιμελητηρίου. Οι εποπτικές αρχές θα ε, ελέγξουν και την εφαρμογή του συστήματος. Ακόμα συζητούμε πώς να εξασφαλίσουμε ώστε αυτές οι δεσμεύσεις πραγματικά να ισχύσουν με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Το δικαστήριο τόνισε ότι μία απόφαση περί επάρκειας θα πρέπει να αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γι' αυτό εργαζόμαστε επί του σημείου αυτού με τις ΕΠΑ έτσι ώστε να γίνεται αναθεώρηση σε ετήσια βάση, με βάση έναν ετήσιο μηχανισμό αναθεώρησης, λαμβάνοντας υπόψη και τις εξαιρέσεις και θέματα εθνικής ασφάλειας. Και αυτό αφορά τις ρυθμιστικές αρχές και από τις δύο πλευρές. Όταν μιλάμε για την παρέμβαση δημοσίων αρχών, ιδιαίτερα για λόγους επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, το δικαστήριο κρίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς όροι και περιορισμοί που να διέπουν το σύστημα. Αυτό αντικατοπτρίζει και τη στάση της Επιτροπής δύο χρόνια πριν. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε με τις ΕΠΑ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να εξασφαλίσουμε επαρκείς περιορισμούς και διασφαλίσεις προστασίας για την προστασία δεδομένων γενικότερα, έτσι ώστε να υπάρχει και νομοθετικός έλεγχος για τις δραστηριότητες αυτές. Να είμαστε απόλυτα σαφείς ως προς το τελευταίο σημείο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της απόφασης του δικαστηρίου, αλλά η συζήτηση, ας μην το ξεχνάμε, ε, γινόταν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μετά τις αποκαλύψεις δύο χρόνια πριν που οδήγησαν και στην υπόθεση και απόφαση του δικαστηρίου, οι ΙΠΑ αναθεωρούν το εθνικό πλαίσιο λειτουργίας ε, του συστήματος πληροφόρησης και πληροφοριών με βάση το Freedom Act και τη την οδηγία 28 του Προέδρου για την εποπτεία και για το γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ατομικά δικαιώματα μη Αμερικανών πολιτών πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερα στοχοθετημένη εποπτεία. Σε σχέση με τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται, επειδή υπήρχε προστασία μόνο σε πολίτες των ΗΠΑ, η προστασία αυτή έχει επεκταθεί και σε Ευρωπαίους πολίτες σε σχέση με τη διάδοση πληροφοριών. Αποτιμούμε αυτές τις ρήτρες διασφάλισης αλλά βλέπω ότι υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία ως προς την εξέλιξη. Επίσης, έχουμε προβάλει μία πρωτοβουλία για νομοθετική προστασία και Ευρωπαίων πολιτών με βάση το Privacy Act των ΗΠΑ. Έχει λοιπόν εγκριθεί αυτό το πλαίσιο από την Βουλή των Κοινοτήτων και θα εγκριθεί και από τη Γερουσία τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα οδηγεί στην περαιτέρω προστασία μεταφοράς δεδομένων. Τώρα θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό και σε άλλα στοιχεία και να αναλύσουμε τις προαπαιτήσεις της απόφασης του δικαστηρίου. Αγαπητά μέλη, κάνω έκκληση στη δική σας δέσμευση και ανάληψη πρωτοβουλίας για αυτή μας την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας μέχρι τώρα στα πλαίσια του θέματος της νομοθετικής αποκατάστασης και θα ήθελα να επεκταθείτε και στους ομολόγους μας της ΕΠΑ, είτε στο Κογκρέσο είτε στη, σε επίπεδο κυβέρνησης. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας και τη βοήθεια των επιχειρήσεων για να πείσουμε της ΕΠΑ ότι χρειάζονται επιπρόσθετα μέτρα. Μια καλή έκβαση είναι πολύ σημαντική για τις ευρύτερες σχέσεις μας με τις ΕΠΑ που είναι ο κύριος στρατηγικός μας εταίρος πολιτικά και οικονομικά. Και όπως σας είπα και πριν, όπως προείπα στην Ολομέλεια, θέλω να υπάρξει ε, σωστή πληροφόρηση για την όλη διαδικασία και σας θεωρώ βασικό μου συνεργάτη. Θα σας ενημερώνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα σταματήσω τώρα για τον ασφαλή λιμένα, για το Safe Harbor και θα ήθελα να σας απαντήσω εάν ε, θέλετε να μιλήσουμε για μια γενικότερη συμφωνία που αφορά τη συνεργασία μας με τη ΣΥΠΑ, μπορώ να σας μιλήσω για τον κανονισμό προστασίας των δεδομένων, αν θέλετε να επεκταθούμε και σε άλλους τομείς της προστασίας. Και όπως είπε και ο Κλοντ, τονίζω ότι προσμένω την ε, επόμενη συνάντησή μας κατά την ε, το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου για να σας ε, μιλήσω για το πρόγραμμα δράσης των ΛΟΑΔ για θέματα όπως η ρίζοσπαστικοποίηση, η καταπολέμηση του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας στην κοινωνία και τη συνεργασία μας με τις επιγραμμικές υπηρεσίες κατά των λόγων μίσους. Και να σας ε, μιλήσω βεβαίως ε, και για το κανονισμό που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. καθώς και τα ευρήματα του Οργανισμού ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε σχέση με τη συμμόρφωση εκεί όπου υπάρχει υψηλή συγκέντρωση προσφύγων στα κράτη-μέλη. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες για την προσεχή συνάντησή μας. Και βεβαίως τα επιμέρους σημεία εξαρτώνται από εσάς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπε. Συνάλφοι, έχουμε περιθώριο μέχρι τις 9 η ώρα. και χωρίς να υποτιμούμε την σημασία του θέματος του ε, ε, ασφαλούς λιμένα ε, αυτός είναι ο χρόνος που έχουμε εννέα ομιλητές έχουν εγγραφεί στον κατάλογο παρακαλώ μην μακρηγορήσετε για να πάρουμε λεπτομερείς απαντήσεις και να αναλύσουμε το, την κατεύθυνση προς την οποία παίρνει το θέμα του ασφαλούς λιμένα. Παρακολουθείτε λοιπόν περιοριστείτε χρονικά για να πάρουμε πλήρες απαντήσεις. Όλοι είναι στον κατάλογο, όλοι όσοι το ζητήσατε. Ε, αν δεν θέλει κανείς άλλος, κρίνω τον κατάλογο. Λόρα Φεράρα ήταν τελευταία. Έχει κλείσει ο κατάλογος τώρα. Ποιος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας επίσης ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που απόψε είσαστε παρούσα να απαντήσετε στις παρατηρήσεις και ερωτήσεις μας γύρω από το θέμα του Safe Harbor, του ασφαλούς λιμένα. Το βρίσκω καλό ότι το προσεγγίζετε ενοιολογικά και έτσι το επεξηγείτε και προχωράτε. Η νομολογία του ΔΕΚ του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είναι καταρχήν σωστή για μας το θεωρώ ίσως ε, όχι τόσο υπεύθυνο το ότι δεν προέβλεψε μεταβατικές περιόδους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ή κάποια πράγματα επί των οποίων θα μπορούσε να βασιστεί κανείς. Ε. Το θεωρώ σωστό ότι τώρα γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθούν ε, νέα θεμέλια ώστε να υπάρξει νομική βεβαιότητα και νομική ασφάλεια. Και γοργά κιόλα επειδή είναι κατεπήγον αυτό. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια κατεύθυνση και γι' αυτό είναι θετικό το ότι εσείς έτσι το προσεγγίσατε όπως μας εκθέσατε. Για τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις προς τη σωστή κατεύθυνση έγιναν μέχρι σήμερα. Με ενδιαφέρει. Έχετε την εντύπωση ότι όλα από την αρχή θα πρέπει να ξαναξεκινήσουν μετά από αυτή την ομολογία, την απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν θα το θεωρούσα εγώ έτσι. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας δεδομένων όταν οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα έχουν το δικαίωμα ιδίας πρωτοβουλίας εξέτασης του αν συνάδουν ή όχι οι διαδικασίες ή όχι. Μήπως εδώ ελοχεύουν κίνδυνοι. Φυσικά θα έπρεπε να υπάρχουν σφαιρικές προδιαγραφές για την προστασία των δεδομένων. Κάτι τέτοιο όμως είναι αυταπάτη αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν να υπήρχαν διατλαντικές τέτοιες προδιαγραφές, ευρωπαϊκές και αμερικανικές. Υπάρχουν όμως ε, ε, δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν αποκλειστικό κριτήριο για την αξιολόγηση ενός αμοιβαίου τέτοιου συστήματος για την προστασία των δεδομένων να ισχύει μια τέτοια ξεχωριστή κατάσταση. Θα, υπάρξει, θα υπάρξουν στεγανά αν δούμε το τι συμβαίνει και στη Ρωσία και στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει επακριβώς να εξετάσουμε και από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διαφορές των νομικών συστημάτων και των νομολογιών. Εγώ πιστεύω βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση για την πιστοποίηση ώστε να υπάρξουν μέτρα ελέγχου τα οποία θα θεσπιστούν και στο τέλος τέλος να μπορεί και η Επιτροπή ίδια να ελέγχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν χαίρομαι για την απόφαση του Ευρωδικαστηρίου. Ταυτόχρονα το βρίσκω όμως κάπως ανησυχητικό το ότι χρειαζόταν ένας φοιτητής να προσφύγει σε ένα δικαστήριο ενώ υπήρχαν επί χρόνια επισημάνσεις και στοιχεία ότι αυτή η συμφωνία δεν δημιουργούσε ασφαλή λιμένα, δεν ήταν ασφαλής λιμένας και όλες αυτές ε, οι ενστάσεις δεν ελήφθησαν, δεν πάθηκαν στα σοβαρά και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι με πολύ βραδείς ρυθμούς ε, υπήρξε πρόοδος και δεν βλέπω και κάποια επιχείρηση να είχε εγκαταλείψει τις δραστηριότητες της λόγω αυτού του, αυτής της απόφασης. Δεν ξέρω γιατί λοιπόν να αναφέρουν κάποιοι ότι κάτι τέτοιο είναι ανεύθυνο. Και στο κάτω-κάτω η απόφαση του δικαστηρίου αφορά και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούμε να πούμε «Α, μέχρι σήμερα δεν ήταν σεβαστά, αλλά συνεχίστε γιατί πρέπει να κερδίσουμε χρήματα και να υπάρξει κέρδος». Δεν έχω όμως πρόβλημα με το ότι οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα έχουν και πάλι ελεγκτικές αρμοδιότητες και δικαιώματα. Εδώ θα, υπάρξουν, ε, θα, στρέψουν το βλέμμα τους με ιδιαίτερη προσοχή να δουν αν υπάρχουν ελλείψεις ή κενά και αυτό είναι θετικό. Όσον αφορά τις εναλλακτικέ λύσεις που ανέφερε η Επίτροπος Γιούροβα, είναι πραγματικά αναγκαίο να καταλήξουμε σε κοινού κανόνες. Διότι <clears throat> αν δεν το κάνουμε αυτό θα καταλήξουμε σε διαφορετικές απόψεις για το τι είναι υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων ή όχι. Και επιτέλους και στο θέμα του ποια συμφωνία θα γίνει με τις ΗΠΑ το θέμα των ελέγχων φυσικά διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά πόσον δηλαδή αρχές προστασίας δεδομένων της Ευρώπης θα μπορούν να ασκήσουν την επιρροή τους για να τηρούνται οι συμπεφωνημένες αρχές και προδιαγραφές. Αλλά εδώ και πάλι δύο διαφορετικά πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Να δούμε τι κάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο, αναβαθμισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων και αφετέρου τι γίνεται με law enforcement, με την επιβολή των νόμων και της νομοθεσίας και τι γίνεται με τις μυστικές υπηρεσίες ποιες αρμοδιότητες και δικαιώματα θα έχουν. Και εδώ διατλαντικά και στη ΣΥΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει πολλά να γίνουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Και όσον αφορά την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα λόγω, ε, μέσω αρχών, κρατικών αρχών επιβολής του νόμου, αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας, πρέπει να είναι η εξαίρεση. Και καταρχήν ε, οι ιδιοκτικές αρχές δεν μπορεί να έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους προσωπικά ιδιωτικά δεδομένα. Mr. Kirkhope, please. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο για τις ε, διευκρινήσεις αρκετών θεμάτων. Θα ήθελα να μου πει τη γνώμη της όμως σε ό,τι αφορά την κατάσταση σήμερα. Ε, σήμερα με την οποία τα δικαστήρια φτάνουν πιο πέρα από την νομοθετική αρχή. Πιστεύει η Κομισιόν ότι το πρόβλημα είναι πιο ευρύ Ε, πολλές φορές οι νομοθέτες θεωρούν ότι κάτι είναι αρκετό, αλλά το, τα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργότερα το κηρύττουν ανεπαρκές. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι όταν συμφωνούμε επί μιας, ενός νομοθετικού κειμένου ε, οι δικαστές δεν θα διαφωνήσουν αργότερα και αυτό να το ξέρουμε εκ των προτέρων. Θα μπορούσε επίσης να μας ενημερώσει για τη σχέση με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Δικαστήριου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι αυτή η απόφαση θα επηρεάσει και άλλες μελλοντικέ διαπραγματεύσεις. Πιστεύετε ότι ε, το γεγονό ότι ε, η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε ε, την νομοθεσία περί επανόρθωσης ε, αποκαθιστά εν το πρόβλημα. Επίσης η Κομισιόν είχε feedback από τις Εθνικές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων των Κρατών Μελών μετά την απόφαση αυτού του δικαστηρίου σε ό,τι αφορά το πώς χειρίζονται αυτοί, αυτές την κατάσταση καθώς επίσης και οι επιχείρησεις τους. Εμείς, ε, μάλλον οι, οι εκλογείς μας, οι φιωφόροι μας έρχονται συχνά σε επαφή μαζί μας και μας ρωτούν, ε, μας ρωτούν αν θα στηριχθούν ε, υπό το φως και εν ώψη μιας καινούριας ε, συμφωνίας ε, και το κατά πόσον, μας ρωτούν το κατά πόσον η σύνεψη μιας τέτοιας ε, καινούριας συμφωνίας θα γίνει με διαφανή τρόπο σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι θα κληθούν να την εφαρμόσουν. Κυρία Ιντβελτ, ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε για την παρουσία σας, για την ξεκάθαρη παρουσίαση της κατάστασης. Έχω πολλές ερωτήσεις όμως. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την ε, δήλωσή σας ότι ο επιχειρηματικό κόσμος χρειάζεται βεβαιότητα, ασφαλώς και επιγόντως, αλλά χρειάζονται, ε, χρειαζόντουσαν ε, βεβαιότητα και τα προηγούμενα χρόνια και εμείς είχαμε ζητήσει την κατάργηση της συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα. Και οι πολίτες επίση χρειάζονται ασφάλεια και βεβαιότητα και οι επιχειρήσεις έχουν κάνει τα στραβά μάτια σε ό,τι αφορά τις αδυναμίες της συμφωνίας ε, περί ασφαλούς λιμένους. Κροκοδίλια δάκρυα λοιπόν. Ε, επίσης, ρωτώ το εξής. Ποια θα είναι πώς θα επηρεάσει αυτή η συμφωνία την, η απόφαση της συμφωνία ομπρέλα τη συμφωνία περί ε, στοιχείων των ε, δεδομένων των επιβατών κλπ. Αυτό είναι πολύ επίγον να το απαντήσουμε. Ε, Υποτίθεται ότι λειτουργούμε, ε, ότι ετοιμάζουμε ε, μια απόφαση για το ε, νέφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ασπίδα προστασίας. Αυτή δεν είναι η λύση. Θέλουμε να είναι ανοιχτό το ίντερνετ αλλά με επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων. Και αυτό με οδηγεί στο θέμα της επιβολής του νόμου. Καταρχήν διάβασα κάπου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δείχνει με το δάχτυλο, αλλά τα προηγούμενα χρόνια μόνο τέσσερις προσφυγές είχαν υποβάλει. Οπότε τι γίνεται με την ε, εφαρμογή των την Κομισιόν. Το άλλο σχετικό θέμα είναι το εξή. Μιλήσατε για τι εθνικέ αρχέ προστασία των δεδομένων. Όπω ξέρω όμω ότι ορισμένε αρχές, ε, γερμανικέ αρχέ κρατηδίων ε, στη Γερμανία είπαν ότι θα αρχίσουμε ήδη από τώρα να εφαρμόζουμε τον νόμο και αν οι επιχειρήσεις, όποιες επιχειρήσεις δεν πληρούν το, το, το πνεύμα του, της ε, συμφωνίας για το ε, ασφαλή ημέρα θα τα βρουν άσχημα. Ε, εδώ, επίση, δεν πρόκειται για διαπραγματεύσει, πρόκειται για μονομερή απόφαση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι, συ, συζητήσει με, ε, με τι Ηνωμένε Πολιτείε οδήγησαν στο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δέχονται πω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάρει μονομερό την απόφαση περί ασφαλού λιμένα, τότε αυτή η απόφαση θα εφαρμοστεί. Αλλά αυτή είναι μια μονομερή απόφαση, δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση. Το έχουμε συζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Τελικά όμως το συμπέρασμα είναι ότι όπως είπε και ο Τίμωθη πιο πριν, εξακολουθούμε και περνάμε και ψηφίζουμε νόμους που τελικά δεν στέκονται στα πόδια τους και μας τους στέλνουν πίσω τα δικαστήρια. Αυτό γίνεται ξανά και ξανά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική συμφωνία που θα αντικαταστήσει τον ασφαλιμένα θα συμμορφώνεται με τα στάνταρ, με τους όρους του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπηρεσίες, ε, μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ από την μια μεριά και οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές υπηρεσίες από την άλλη μεριά και όπως ε, λέτε πολύ σωστά όλες όλες έχουν υπερβεί τα όρια τους και τα καθήκοντά τους, πώς αυτές οι δύο θα ε, αναγκαστούν να συμμορφωθούν με, τα, με τους όρους, με τους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Είναι σημαντικό ήρεμα νυφάλια να ανταλλάξουμε απόψεις και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Αμέσως περνάω στην ουσία του θέματος. Η πρώτη ερώτηση προς εμάς είναι είπατε ότι θέλετε μία δήλωση να εγκρίνετε με συγκεκριμένα σημεία κέντρου βάρους τι θα γίνει με τις επιχειρήσεις. Πώς φαντάζεστε μια τέτοια δήλωση, ποια θα είναι τα σημεία πυρήνες, τα κύρια σημεία αυτής της δήλωσης για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε πραγματικά η ερμηνεία της ε, απόφασης του ΔΕΚ να μπορεί να ενταθεί σωστά, ώστε να υπάρξει νομική βεβαιότητα για αυτές τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, με εκπλήσει όλο και περισσότερο ότι εκατό φορές αποτύχαμε και είδαμε αυτή την αποτυχία ενώπιόν μας σαν την καταβήθηση του Τιτανικού και δεν χρειαζόταν η νομολογία του 10 ξέραμε ότι αυτό δεν λειτουργούσε και γίνεται διαρκώς η προσπάθεια να υπάρξει ο ασφαλής λιμένας. Ερωτώ πώς θα τα καταφέρετε μια και ε, διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι τα προσωπικά δεδομένα ακόμα και με καταπληκτικούς ελέγχους των ε, αρχών προστασίας και στη ΣΥΠΑ όμως με την πρόσβαση που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποτυγχάνει το εγχείρημα και δεν είναι αίσιος ο λιμένας, δεν είναι ασφαλής ο λιμένας. Τι είδου λοιπόν απόψεις έχετε για τον ασφαλή λιμένα. Αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Πώς θα αντιμετωπίσετε το κύριο πρόβλημα της εθνικής ασφάλειας ε, στα κράτη-μέλη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Καταλήγουν τα στοιχεία αυτά στις μυστικές υπηρεσίες, άσχετα ποιοι έλεγχοι γίνονται και ποιος ασφαλής λιμένας ισχύει εκ περιτροπής. Πώς θα υπάρξει, πώς θα διαμορφωθεί το σύστημα ελέγχων και πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια adequacy position, μια τέτοια επαρκής για την ασφάλεια κατάσταση και το τελευταίο σημείο, σημείο φυσικά είναι οι επιπτώσεις. Έχουμε SWIFT, έχουμε όλα αυτά τα πλαίσια στα οποία λειτουργούν τα θέματα προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει όμως σαφήνεια το τι σημαίνουν όλα αυτά. Παρακαλώ θερμά να μας πείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα υπάρξουν και να αποσαφινιστεί αυτό. Και ελπίζω ότι θα είναι τόσο θετική η προστασία των δεδομένων μέσω της νέας ρύθμισης ώστε να είναι αποτελεσματική. Ευχαριστώ. Thank Άλμπρεχτ παρακαλώ. Ευχαριστώ Επίτροπε για το ότι επεξηγήσατε τις απόψεις σας ε, σε σχέση με την απόφαση του ΔΕΚ ε, ακούγοντας ε, τις θέσεις αυτές και με τις ερωτήσεις αυτές η πρώτη μου παρατήρηση και ερώτηση θα ήταν σε σχέση με το σήμερα τώρα, δίνοντας συνέχεια σε μια νέα ρύθμιση και σε μια νέα ρύθμιση για την επάρκεια. Διαρωτώ με πραγματικά όμως, επανειλημμένα διαρκώς από την ομολογία του ΔΕΚ, πώς επιθυμείτε να προσαρμόσετε μια νέα απόφαση, δηλαδή να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του δικαστηρίου, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση και δεν είσαστε σε θέση να το κάνετε αυτό, να αλλάξετε δηλαδή το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη ΣΥΠΑ και μάλιστα εντός ε, ε, και μάλιστα προσεχώς. Είναι σαφές το 10 ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΠΑ δεν επιτρέπουν για ένα αναγκαίο αντιστάθμισμα, αμοιβαίο αντιστάθμισμα για την επαρκή προστασία. Για τι πράγμα συζητούμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ρυθμιστούν αυτά τα θέματα έγκαιρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δεν νομίζω λοιπόν. Απλώς ερώτηση υποβάλλω. Θα ήθελα να έχω επεξηγήσει από πλευρά σας, περαιτέρω ερμηνείες για το πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτό το αίτημα. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Πώς θα ανταποκριθείτε στα μελήματα, στις ανησυχίες του δικαστηρίου. Και το επόμενο ερώτημα. Γιατί. Διότι τώρα το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο των ΙΠΑ. Και αν ΙΠΑ επιθυμούν οι επιχειρήσεις τους να έχουν μια ρύθμιση ως μια ρύθμιση επάρκειας που θα είναι προνομιακή πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές μια και οι άλλοι δεν θα έχουν μια τέτοια πιστοποίηση επάρκειας δηλαδή δεν θα είναι δυνατόν να υπάρχει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά με άλλο τρόπο γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε αυτό το θέμα τώρα να το αντιμετωπίσει με αυτόν τον τρόπο, Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να ρυθμίσει αυτό το θέμα. Οι εταιρείε του να προσεγγίσουν την κυβέρνηση των ΗΠΑ ώστε να υπάρξει αναγκαία προσαρμογή. Απλώ ερώτηση υποβάλλω για να μα επεξηγήσετε τα σχετικά. Και κάνουμε και λόγο φυσικά για το σεβασμό σε αυτή την απόφαση του ΔΕΚ. Και είναι απόλυτα σωστό η ερώτηση του Τίμωθη Κέρκοπ Πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρξει άλλη απόφαση του δικαστηρίου. Να μην υπάρξει δηλαδή νέα διαπίστωση παραβίασης ε, του νομικού πλαισίου και να χρειάζεται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε ένας πολίτης να προσφύγει με δική του προσφυγή στο 10 ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση. Και πώς θα τα ρυθμίσει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δική της πρωτοβουλία Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. Αλλά δυστυχώ χρειάζομαι άλλο ένα λεπτό γιατί θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα άλλο σημείο που είναι πιστεύω και αυτό σημαντικό. Αναφέρθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στι αποκαλύψει του Έντουαρντ Σνόντεν σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία είχε παρακολουθήσει και την ε, ανάμειξη των μυστικών ε, υπηρεσιών. Είπε το δικαστήριο πρώτον οι αποκαλύψεις αυτές είναι ουσιαστικά αληθείς και τις λαμβάνουμε υπόψη σοβαρά και είναι ένα θέμα <clears throat> για την ε, ε, εποπτεία αυτών των θεμάτων. Αν συμβαίνει αυτό θα ήθελα να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επ' αυτού. Δηλαδή κάποιο τμήμα αυτών των αποκαλύψεων αφορά τα δικά μας κράτη-μέλη και το επίπεδο των θεμάτων ε, εθνικής ασφάλειας και την παραβίαση αρχών, αρχών που αφορούν την ασφάλεια αυτών των δεδομένων. Γιατί δεν ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασίες ε, επιπροσφυγή εις βάρος εκείνων των κρατών μελών που ξεπερνούν τα εσκαμμένα όσον αφορά τον τομέα της εθνικής ασφάλειας και το τι θα έπρεπε να καλύπτεται από τη νέα νομοθεσία, νέα νομολογία και τι θα έπρεπε να εντάσσεται στην προστασία των θεμελιωδών δεδομένων από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα θέματα εθνικής ασφάλειας να είναι κατανοητά και σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών και η προστασία των δεδομένων σε σχέση με την ομολογία. Λοιπόν, και ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρεται στην απόφαση αυτή. Σε σχέση δηλαδή με την οδηγία αποθήκευσης ε, των προσωπικών δεδομένων που πάλι εδώ η μαζική ε, ε, παρακολούθηση και ανάμιξη των αρχών κατασκοπίας των μυστικών υπηρεσιών στα προσωπικά δεδομένα τα κράτη-μέλη έχουν αυτά τα μέτρα που ισχύουν. Θα πρέπει να επιβληθεί λοιπόν αυτή η νομολογία έναντι των κρατών μελών και να, να σεβαστούν τα κράτη-μέλη αυτές τις αρχές. Η κυρία Φεράρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση σήμερα γιατί η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί πλήγμα στις, ε, γιατί είπα και το σύστημα πληροφόρησης και εποπτείας τους, γιατί ε, δυστυχώς αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η κατασκοπία κατά των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων. Γι' αυτό και θα πρέπει ε, πολλές φορές να περιορίζονται οι εθνικές επεμβάσεις Χρειάζεται μία λύση ώστε να αλλάξει ο Αμερικανικός νόμος. Όχι ενημέρωση του παρόντος συστήματος του Safe Harbor. Αναρωτιόμαστε τι θα κάνει η Επιτροπή. Θα περιοριστεί στην ενημέρωση ή θα προβεί σε νέα συμφωνία και πώς θα διασφαλίσει την τήρηση της απόφασης του δικαστηρίου το Safe Harbor θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στις διατλαντικές συναλλαγές. Πώς ε, θα διαχειριστεί η Επιτροπή τη μεταβατική περίοδο και τι θα γίνει εάν οι επιχειρήσεις αλλάξουν τη συμφωνία τους με τους Ευρωπαίους χρήστες, έτσι ώστε να αλλάξει το, το πνεύμα της προστασίας δεδομένων στο εξωτερικό. Ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις και τέλος, τα κράτη-μέλη μπορούν να αναβάλουν τη μεταφορά δεδομένων προς τις ΗΠΑ και να ζητήσουν να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο ευρωπαϊκό έδαφος. Ίσως ε, αυτό θα ήταν ένα ενδεχόμενο σενάριο. Μπορείτε να το επαληθεύσετε. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πόνη; Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε που βρίσκεστε εδώ. Νομίζω ότι η συζήτηση είναι ύψη της σημασίας γιατί τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κήρυξε άκυρη τη συμφωνία περί ασφαλούς λιμένα, θα πρέπει να δούμε όχι μόνο τη μεταφορά δεδομένων προς τη ΣΥΠΑ, αλλά και τις ε, συνέπειες ως προς τη συμφωνίες επάρκειας για την προστασία δεδομένων. Συμφωνώντας με πολλές δηλώσεις σήμερα, θα ήθελα να υποβάλω τρία ερωτήματα. Η μεταφορά σε τρίτες χώρες αφορά αποφάσεις επάρκειας σε σχέση με τις συμβατικές ρήτρες και το εταιρικό δίκαιο. Και αυτό αναπερίπτωση σύμφωνα με τις ε, κρατικές αρχές. Αυτά ως προς την ε, μεταβατική περίοδο. Αυτό όμω αρκεί αν λάβουμε υπόψη την εργασία του Αμερικανικού Κογκρέσου γιατί μέσα στα πλαίσια της επάρκειας και της αντιστήχησης θα προβάλλεται ένα νέο πλαίσιο εργασίας για αυτές τις σχέσεις. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ορισμένα από τα μέσα που προανέφερα χρησιμοποιούνται από μεγάλες επιχειρήσεις, όχι μικρές τι λύσεις μπορούμε να προβάλλουμε για τις ΜΜΕ, τι υποστήριξη δηλαδή από τις αρχές προστασίας των δεδομένων. Τι σημαίνει αυτή η απόφαση για το, για το γενικότερο σύστημα επάρκειας. Πώς θα πρέπει να γίνουν κατανοητές αυτές οι αποφάσεις από τις επιχειρήσεις. Και τέλος, οι οργανισμοί προστασίας δεδομένων πώς ε, θα πρέπει να κατανοήσουν αυτή την απόφαση. Το Δεκέμβριο βεβαίως θα προβάλλουμε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το βρίσκω και εγώ πολύ θετικό το ότι κάνατε την προσπάθεια με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να τοποθετηθείτε και να εξετάσετε τα θέματα των επιχειρήσεων σε αυτό το εγχείρημα. Έχω μια έννοια που αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και δεν βλέπω εδώ να αναφέρεται κάτι σχετικά και έχω τον φόβο ότι το σύνολο είναι μια επανόρθωση, μια διορθωτική δράση και δεν έχει ε, δράση, ε, δεν είναι δράση επιθεμάτων αρχής και το ζήτημα το ότι τα νομοθετήματα, οι νόμοι δεν είναι τόσο καλοί, δεν είναι τόσο θετικοί στο αποτέλεσμά τους ώστε να υπάρχουν προσφυγές στο 10 τότε δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλά για better regulation, regulation καλύτερη νομοθεσία, αλλά θα έπρεπε να είναι πιο αποτελεσματική στη σύνταξη των νομοθετικών προτάσεων για να γλιτώσουμε όλη αυτή τη φασαρία. Τρεις σύντομες ερωτήσεις με βάση την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου διαπιστώνεται ότι η νομολογία στις ΗΠΑ ε, στον πυρήνα των θεμάτων προστασία δηλαδή προσωπικών δεδομένων δεν υλοποιεί σε πλήρη βαθμό τις απαιτήσεις. Και τώρα ένας ασφαλής λιμένας Safe Harbor 2 δεύτερος δηλαδή δεν θα σήμαινε μια μεταρρύθμιση εκβάθρων του νομοθετικού πλαισίου των ΗΠΑ. Είναι όμως κάτι τέτοιο ρεαλιστικό Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Διαπίστωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η προστασία πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το ζήτημα, το εκάστοτε ζήτημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια θέματα θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλότερο επίπεδο, αναβαθμισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σχέση με το σήμερα. Τρίτον, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ε, την ε, ρήτρα, πάγια ρήτρα επί των αρχών, στερεότυπα. Το βρίσκω θετικό, όμως σε σχέση με τις επιχειρήσεις, την εξαίρεση σε σχέση με το άρθρο το σχετικό άρθρο δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή των όρων. Πώς το βλέπετε αυτό. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, διότι νομίζω είναι ένα γενικότερο θέμα αυτό. Ποιο χρόνο απαιτεί κάτι τέτοιο, ποιο χρόνο ορίζοντα θα προβλέπατε εσείς. Ευχαριστώ. Mr. Le Breton, please. Le Breton, παρακαλώ. Madame la Commissaire. Κύριε Επιτροπέ, είναι πολύ σημαντικό σήμερα να γίνει μια συζήτηση για την απόφαση του Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχει το θετικό ότι προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ιδιαίτερο τα ατομικά, τα προσωπικά δεδομένα. Από αυτή την έννοια είναι κρίσιμο, κρίσιμη αυτή η απόφαση, ε, ιστορική. Και ως μέλος της Επιτροπής ε, το υπογραμμίζω αυτό. Το βασικό όμως ενδιαφέρον δεν είναι αυτό, είναι ότι καταδικάζει διπλά ε, τις ε, της Κομισιόν, της οποίας είστε μέλος. Προσπαθείτε βέβαια να ελαχιστοποιήσετε το βεληνικές αυτής της απόφασης, αλλά δεν πείθετε. Λέτε ότι χρειάζεται ένα καινούργιο πλαίσιο προστασία των δεδομένων στι ανταλλαγέ με τι ΟΠΑ και υπογραμμίζεται ότι πρέπει οι εθνικέ αρχέ προστασία δεδομένων να παίξουν ένα πιο ε, δυναμικό ρόλο. Ε, καλά κάνετε και το λέτε, <laughs> αλλά ε, διότι βέβαια αυτό που πρώτα πρώτα λέει η απόφαση είναι ότι δείχνει η Κομισιόν να έχει υπερβολικές εξουσίες, κάτι που έχει περιορίσει υπερβολικά με τη σειρά του τις αρμοδιότητες των εθνικών ε, ε αρχών προστασίας δεδομένων, οπότε πολύ σωστά βέβαια λέτε ότι πρέπει να ε, γίνουν σεβαστές αυτές οι αρχές. Δεύτερον, λέτε ότι δεν αξιολογεί το αμερικανικό σύστημα αυτή η απόφαση, πολύ διπλωματική η, δήλωσή σας. Το αντίθετο συμβαίνει. Το, η απόφαση αυτού του δικαστηρίου είναι πολύ αυστηρή για το αμερικανικό σύστημα. Γιατί, γιατί το σύστημα πρώτον δεν προστατεύει επαρκώς τα προσωπικά δεδομένα και δεύτερον διότι το χαμηλό επίπεδο προστασίας δεν εφαρμόζεται καν στους Ευρωπαίους πολίτες. Οπότε λέτε ότι θα πρέπει να υποχρεώσουμε τους ε, εταίρους μεσοαμερικανούς να βελτιωθούν και ότι μπορεί ενδεχομένω να τροποποιηθούν ή να πρωτοποθηθεί η να η νομοθεσια τους περί ιδιωτικής ζωής κλπ. Αλλά ε, από ό,τι πιστεύω εγώ δεν πρόκειται να τα καταφέρετε διότι ε, οι Αμερικάνοι έχουν ε, μια αρετή προστατεύουν τα συμφέροντά τους και δεν είναι διαλλακτικοί όταν πλήττονται αυτά τα εθνικά συμφέροντα. Η Κομισιόν έδειξε ότι είναι αδύναμη διότι, έχει, διότι κατά βάση τι έκανε, θυσίασε το επίπεδο προστασίας των, ε, ατομικών δικαιωμάτων ε, προκειμένου στο βωμό μάλλον της υπογραφής αυτής της συμφωνίας. Ε, από ό,τι φαίνεται οι επιχειρήσεις υπερτερούν έναν της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ευχαριστώ. Ο κ. Λόπες Αγγιλάρ. Commissioner, Commissioner ε, Επίτροπε, και εγώ πιστεύω ότι αυτή η απόφαση του Δικαστήριου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, είναι ιστορική σημασίας ε, και θα διαμορφώσει την κουλτούρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιώδων δικαιωμάτων και τις μελλοντικές ερμηνείες όλων των νομοθετημάτων, σχετικών νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα αναμενόμενο και των συμφωνιών με τρίτες χώρες. Το πρόβλημα είναι ότι εστιάσαμε υπερβολικά στο πρόγραμμα ασφαλούς λιμανά με τις ΗΠΑ ενώ η απόφαση αυτή έχει πολύ μεγαλύτερο βεληνικές. Ε, επηρεάζει τις διμερείς συμφωνίες με οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αξιολογείτε τις συνέπειες αυτή αυτής της απόφασης, όχι μόνο σε αυτή τη συμφωνία, αλλά και σε άλλες συμφωνίες που περιλαμβάνουν κεφάλαια ε, μεταφοράς ε, προσωπικών δεδομένων. Για παράδειγμα, η TGIP που έχει σχέση με πρότυπα προστασία, με κάνω προστασία προσωπικών δικαιωμάτων. Επίση, τι επιπτώσει έχει αυτή η απόφαση ε, στι εσωτερικέ παρακολουθήσει ε, των πολιτών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των κρατών μελών. Θα ήθελα να μου πείτε την εκτίμησή σας και για αυτό το θέμα. Επίση, αναφέρατε και άλλε φιλοδοξίε που έχετε να σας πω το εξής σε ό,τι αφορά την πρόθεση ε, της αντιμετώπισης του, του θέματος των, ε, του, των δηλώσεων ε, και σχολείων μίσους ε, στο διαδίκτυο. Ε, αυτό ξεπερνάει τη συμφωνία πλαίσιο. Ε, αυτό που μας είπατε ξεπερνάει τη συμφωνία πλαίσιο και θέλω να πείτε την εκτιμήσή σας. Ευχαριστώ και ο Στίβενς. de tussen Ευχαριστώ πολύ. Κατά την περίοδο μεταξύ της απόφασης του δικαστηρίου και της έγκρισης μιας νέας συμφωνίας, η προστασία των ε, πολιτών είναι χαμηλότερη από ποτέ. Φτάνουμε σε ένα εθνικό κατακαιρματισμένο σύστημα όπου κάθε κράτος προβάλλει το δικό του σύστημα η Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίσει τις διαφορές που υπάρχουν στις ε, διαφορετικές νομοθεσίες όπως ε, την οδηγία για την παρακράτηση των δεδομένων. Δεν θα πρέπει να καταστεί ενεργή αυτή η οδηγία. Δεν ξέρω πώς οι ΜΜΕ θα ασχοληθούν με αυτό το σύστημα. Πιστεύω ότι θα φυγούν με τις γραφειοκρατικές, από τα γραφειοκρατικά μάλλον παρακλάδια αυτής της απόφασης. Τι θα γίνει με τις ΜΜΕ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ Επίτροπε που είστε εδώ. Πολλές φορές η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλήττεται από τον ευρέως διαδεδομένο λαϊκισμό και ίσως οι αποφάσεις του δικαστηρίου να μας καθοδηγήσουν έτσι ώστε να προστατεύσουμε τους πολίτες με συγκεκριμένες δράσεις. Δεν θα ήθελα να ε, επαναλάβω τις ερωτήσεις των προλαλισάντων, απλώς θα εντείνω το περιεχόμενό τους. Πώς θεωρείτε ότι η απόφαση αυτή θα επηρεάσει τον διάλογο μεταξύ Ευρώπης ε, Αμερικής σε σχέση με τη συμφωνία Τίζα και TTIP, σε σχέση με την ανταλλαγή ε, πληροφοριών. Ευχαριστώ. Άννα, είχα κλείσει τον κατάλογο, γι' αυτό δεν θα ήθελα να επεκταθείς πάνω του ενός λεπτού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, Επίτροπε, κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου έχει επιπτώσει στη γενικότερη συμφωνία Umbrella Agreement και σε σχέση με το TTIP, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Πριν δώσω το λόγο στην Επίτροπο, με, θα ήθελα να πω ότι μετά την απόφαση για την παρακράτηση προσωπικών δεδομένων δεν ε, ε, ανέκυψαν άλλες ανακοινώσεις και γι' αυτό έχετε θίξει το θέμα για τις επιπτώσεις στο TTIP και την ε, προστασία των δεδομένων. Είδα, ε, κύριε Επίτροπε, ότι κρατάτε, κρατήσατε πολλές σημειώσεις. Υπάρχει το θέμα που έφυξε όμως και ο κύριος Άλμπρεχτ για, το, για τις ευθύνες των Αμερικανών και θα ήθελα και εγώ να κάνω μία πρόταση και να πω ότι εμείς ως ε, Κοινοβούλιο δεν αντιδράσαμε ε, για κάποιο χρονοδιάγραμμα. Ως προς τις αποφάσεις για τον ασφαλή λιμένα, οι δικαστές ήξεραν τι, ήξεραν τι έκαναν. Όπως είπε ο κύριος Κέρκοπ, ήξεραν ότι δημιουργούν πάγια νομολογία οι δικαστές, ότι διαμορφώνουν τον νόμο, ήξεραν ακριβώς τι κάνουν και γι' αυτό χρειαζόμαστε μία ανακοίνωση της Επιτροπής σε σχέση με τις συνέπειες της απόφασης μέχρι το Δεκέμβριο, ίσως για να δούμε πώς ε, θα διαμορφωθούν οι συμβατικές ρήτρες, πώς θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις οι επιπτώσεις για τις συμφωνίες PNR και TTIP. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Θα πρότεινα λοιπόν μία ανακοίνωση από την Επιτροπή μέχρι το Δεκέμβριο. Γιατί έχει σημασία να δούμε πώς ε, ε, θα διαμορφωθούν και οι συζητήσεις σας με τη ΣΥΠΑ. Γιατί δεν έχουμε παρκή στοιχεία και χρειαζόμαστε να έχουμε περισσότερα στοιχεία πριν από τις συζητήσεις ε, με τη ΣΥΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να λάβετε το λόγο, κυρία Επίτρεπε, για να απαντήσετε ως των δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Να ζητήσω συγγνώμη καταρχήν, διότι ενδεχομένως δεν σημείωσα όλες τις ερωτήσεις. Ελπίζω οι συναδελφοί μου να μου επιστήσουν την προσοχή αν ξεχάσω κάτι. Και Πώς καταρχήν. Και Βος, συγγνώμη. Μίλησε για τις προσεγγίσεις των κρατών μελών και τις εθνικές ε, αρχές προστασίας των δεδομένων και άλλες ερωτήσεις. Ίσως θα ήταν καλύτερα λοιπόν να ξεκινήσω με τη δική μου αξιολόγηση για την σημασία της απόφασης αυτής. Το γεγονός ότι ένα άτομο αντιλαμβάνεται ότι ε, έχουν τύχει παραβίαση τα προσωπικά ατομικά δικαιώματα και μπορεί να πάει στο δικαστήριο και να δικαιωθεί αποτελεί κατά την άποψή μου ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου ότι λειτουργεί το σύστημα θεωρώ ότι η απόφαση αυτή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα σημαντικό βήμα που θα μας βοηθήσει να ολοκληρώσουμε επιτυχώς τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ γιατί δίνει καλύτερους ε, ορισμούς, δίνει καλύτερο ορισμό του τι σημαίνει η επάρκεια. Ε, διαπραγματευόμαστε την συμμόρφωση με τις 13 ε, συστάσεις που εκδόθηκαν το 2013. Ο κ. Βος ρώτησε αν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Όχι δεν θα ξεκινήσουμε ξανά από το μηδέν στις διαπραγματεύσεις μας. Θα χρησιμοποιήσουμε, χρησιμοποιούμε τι, τα επιτεύγματα που είχαμε εξασφαλίσει. Θυμάστε ότι τον Αύγουστο σταματήσαμε τις διαπραγματεύσεις παρόλο ότι είχαμε πετύχει πολλά στις συστάσεις 1 ως 11 που αφορούσαν την συνεχή παρακολούθηση και εφαρμογή αυτού που εγώ ονομάζω εμπορικό κομμάτι. Σταμάτησα όμως οι διαπραγματεύσεις και οι Αμερικάνοι ε, ομόλογοι γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι απαντήσεις που παίρναμε και περιμέναμε από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβριο να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Από σεβασμό προς το δικαστήριο. Θέλαμε πρώτα να ακούσουμε τη γνώμη του δικαστηρίου για την αξιολόγηση της επάρκειας και είμαι πεπισμένη ότι πράξαμε σωστά που περιμέναμε και δεν τελειώσαμε, δεν οριστικοποιήσαμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων το καλοκαίρι. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν λοιπόν. Ε, δεν ε, έχουμε πλησιάσει πολύ στην, ε, στην επίθεση Το αποτέλεσμα κοινών στάνταρ, κοινών προτύπων, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα επιτευχθεί και αυτό. Οι Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ θα πρέπει να έχουν κοινά πρότυπα προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Θέλω όμως να απορρίψω ε, ομά. Ε, αυτό που είπε κάποιος ότι θυσιάσαμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στο βωμό των επιχειρήσεων. Δεν ισχύει αυτό. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, είναι πολύ ψηλά στην εκτίμησή μας και το επίκεντρο των προσπαθειών μας, όχι μόνο στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, αλλά και με άλλες χώρες. Διαπραγματεύσεις για την μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων και άλλα κεφάλαια είναι στο επίκεντρο τέτοιων συμφωνιών, τέτοιων διαπραγματεύσεων. Ε, το ασφαλής λιμένας θα, καθορίζει καλύτερα τη διαδικασία επιστοποίησης, τους μηχανισμούς ελέγχου, ε, τους εξοφίτσιο ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται και τις ε, ε, κυρώσεις που θα πρέπει να επιβάλλει η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου καθώς επίσης θα περιλαμβάνει και μια πολύ σαφή ε, ένα πολύ σαφή προσδιορισμό των εξαιρέσεων διότι μιλήσατε και εσείς για εξαιρέσεις και τους περιορισμούς με βάση τους οποίους οι υπηρεσίες πληροφοριών θα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με το πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα. Το είπα και πριν από έξι μήνες, <laughs> αλλά εξακολουθεί να παραμένει στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να έχουμε σαφή όρια, μια σαφή περιγραφή, καθώς επίσης και τους μηχανισμούς ελέγχου ε, ότι αυτά τα σαφή όρια την χάνουν σεβασμού. Και το είπα και στην εισαγωγική μου ομιλία σήμερα. Ο συνεχής έλεγχος θα διενεργείται ε, και μέσω ετήσιων εκθέσεων από τις Εθνικές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων και θέλουμε η ετήσια ε, και οι επιχειρήσεις να κάνουν και οι ίδιες ετήσιες εκθέσεις. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία ακόμα διαπραγματευόμαστε το κατά πόσον α, τέτοιου είδους επιχειρηματικές αιτήσει εκθέσεις θα είναι υποχρεωτικές ή όχι. Εμείς πιέζουμε προκειμένου αυτές οι εκθέσεις να γίνουν υποχρεωτικές και όχι προαιρετικές. Ακριβώς διότι χρειαζόμαστε σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των περιπτώσεων, ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ε, συναντήθηκα με τους εκπροσώπους του Αμερικανικού ε, Εμπορικού Επιμελητηρίου και με τις Αμερικανικές επιχειρήσεις και διαπίστωσα, ή μάλλον το πω αλλιώ, είδα ότι αντέδρασαν θετικά ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της υποβολής εκθέσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων. Όμως δεν μπορώ να πω κάτι οριστικό για αυτό το ζήτημα. Κυρία ΣΥΠΑΣ σε ό,τι αφορά τις ανατικές λύσεις ε, για τις επιχειρήσεις και πώς θα τις χειριστούμε. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, διότι πλέον επικρατεί νομική αβεβαιότητα και για τις μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και για τις μικρότερες. Όταν, Όταν μιλώ με επιχειρήσεις πάντοτε Επιμένω ότι οι συμμορφούμενες με τους όρους του ασφαλούς λιμένα ε, έπραταν πάντοτε καλή την πίστη. Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να βρούμε μια βιώσιμη λύση το συντομότερο δυνατό. Εγώ αυτή την βλέπω, αυτή τη λύση τη βλέπω σε ένα πιο ασφαλές πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα. Εν τω μεταξύ θα προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις. Τώρα βέβαια αυτό επαφίεται περισσότερο στις αρχές προστασίας των δεδομένων που θα είναι αυτές οι οποίες από εδώ και πέρα θα εφαρμόζουν όχι μόνο την νομοθεσία αλλά και την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξηγούμε σε επιχειρήσεις ότι υπάρχουν εναλλακτικέ έναντι του ασφαλούς λιμένα, διότι εμείς το πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα το θεωρούμε, ότι, το θεωρούμε ως ένα ιδιαίτερο, ειδικό πρόγραμμα για τα δεδομένα τα οποία μεταφέρουν τις ΗΠΑ. Όταν συγκρίνω αυτές τις αναλλακτικέ λύσεις, τις οποίες ήδη σας παρουσίασα. Παράδειγμα, ε, ε, ε ενοχικοί κανόνες, ε, συμβατικοί κανόνες, συγγνώμη, και άλλες αναλλακτικέ λύσεις, όταν τις συγκρίνουμε, διαπιστώνουμε ότι η προστασία θα είναι χαμηλότερη από αυτή που θα είχαμε αν ενισχύαμε το καθεστώς ε, ασφαλούς λιμένα μετά από ε, διαπραγματεύσεις. Τώρα οι επιχειρήσεις χρειάζονται σαφείς οδηγίες και θα τις εκδώσουμε αρχές Νοέμβρη. Χρειάζονται επίσης ε, ενοποιημένους κανόνες και αυτό είναι σημαντικό, το συζητήσαμε με την ε, ομάδα εργασία του άρθρου 29 όπου εκπροσωπούνται οι Εθνικές Αρχές Προστασίας των Δεδομένων. Από τη συνάντηση μαζί τους αντελήφθην ότι και οι ίδιες καταλαβαίνουν πως μια ενιαία προσέγγιση θα βοηθήσει προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτή την ενδιάμεση δύσκολη περίοδο και να διευκολύνουμε τις εταιρείες. Ε, μίλησα τηλεφωνικά και με την κυρία Πρίτσκα που είναι η ε, Αμερικανίδα υπουργό, η οποία μου επανέλαβε ότι και η Αμερικανική πλευρά επιθυμεί μια ενιαία προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή 28 νομικά συστήματα σε 28 κράτη-μέλη. Γι' αυτό το λόγο βιαζόμαστε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, μεταρρύθμισης του, της προστασίας των δεδομένων που θα αντικαταστήσει αυτά τα 28 εθνικά συστήματα και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα. Να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να λάβουν έγκαιρα πληροφόρηση και σαφείς οδηγίες δεν σημαίνει ότι θυσιάζουμε τα ανθρώπινα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Να το υπογραμμίσω μία ακόμα φορά. Κύριος Κίρκοπ μίλησε για το, ρώτησε, για το πώς βλέπουμε τη σημερινή κατάσταση, πώς θα βρούμε κοινά στάνταρ, προδιαγραφές, όρους. Η απάντηση είναι σαφής. Πρέπει να εφαρμόσουμε και να σεβαστούμε την απόφαση του ε, δικαστηρίου που θα αποτελέσει πλέον το πλαίσιο για την αξιολόγηση της ε, επάρκειας. Και οι διαπραγματεύσεις για το νέο πρόγραμμα ασφαλούς λιμένα θα πρέπει να γίνουν κατανοώντας πολύ καλά καταρχήν τις απαιτήσεις του δικαστηρίου. Γι' αυτό το λόγο κάναμε μια πολύ λεπτομερή ανάλυση του τι έχουμε πετύχει μέχρι τώρα στις διαπραγματεύσεις για τον ασφαλή λιμένα. Ποιες είναι οι καινούριε απαιτήσει του δικαστηρίου και τι είναι εφικτό να γίνει. Ορισμένοι από εσά το είπατε ήδη, βέβαια, το είπα και εγώ στην αρχή, ότι ε, το, το πιο δύσκολο, τα πιο δύσκολα κομμάτια είναι αυτά τα οποία επηρεάζουν την αμερικανική νομική τάξη αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο τις νομοθετικές πράξεις ε, που έχουν υιοθετηθεί από το Κογκρέσο, αλλά και ε, αποφάσεις της εκτελεστικής εξουσίας. Γι' αυτό το λόγο διαπραγματευθήκαμε με το Υπουργείο Εμπορίου ε, ε, λύσεις ε, οι οποίες δεν θα, χρεια... απαιτούσουν από εμά να περιμένουμε αλλαγές της ε, ε, αμερικανικής νομοθεσίας. Αυτές θα πάρουν πολλά χρόνια. Χρειαζόμαστε μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα αποφάσεις σε εκτελεστικό επίπεδο. Και βέβαια μακροπρόθεσμα περιμένουμε ε, πιο συνολική και πιο βαθιά μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασία των προσωπικών δεδομένων στι ΗΠΑ. Κάτι όμω που δεν περνάει από το χέρι μα. Γιατί έτσι κι αλλιώ αυτό που διακυβεύεται είναι η εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε οι Αμερικανοί εταίροι μας να καταλάβουν καλύτερα ποια είναι, ποιες είναι οι δικές μας προδιαγραφές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτό όμως είναι κάτι που θα πάρει αρκετό χρόνο. Αρκετοί από εσά μιλήσατε για τις επιπτώσεις του TTIP και του PNR, αλλά και μία ερώτηση υποβλήθηκε. Κυρία Σίπελ, γιατί δεν αναστήλαμε ε, το πλαίσιο αυτό, δηλαδή τη, γιατί να στείλαμε το όλο πλαίσιο και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί πολλοί λέτε ότι δεν υπάρχει επαρκής ε, ε, προστασία από την Αμερικανική πλευρά, άρα ας αναστείλουμε και τον ασφαλή λιμένα. Για μένα αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο Παράλληλα, ε, είχα πολλές σκέψεις γιατί αν αναστείλουμε το Safe Harbor, ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Υπάρχει σχέδιο Β. Αυτό κάνουμε τώρα για μια μεταβατική λύση, αυτό το σχέδιο Β. Η οδηγία έχει τεθεί ενισχύ και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εναλλακτικά μέτρα τα οποία σας προανέφερα. Πριν ε, επεκταθώ στο TTIP θα ήθελα να πω ότι κάποιος υπέβαλε την ερώτηση για τις ε, δυνατότητες των ε, εποπτικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων γιατί τώρα έχουν μεγαλύτερο έργο μεγαλύτερο μερίδιο ας το πούμε έτσι της εργασίας για τη θέση σε ισχύ για την επιβολή μάλλον. Γι' αυτό θεωρώ ότι η ενίσχυση των εξουσιών των εποπτικών αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων ε, είναι ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να ε, ληφθεί μέσα στα πλαίσια της γενικότερης μεταρρύθμισης προστασίας των δεδομένων. Αφού εγκριθεί θα έχουμε δύο χρόνια για πραγματική ειδική προετοιμασία επιχειρησιακής ε, εργασίας που θα υποβάλουμε στους εταίρους για την, τον κανονισμό προστασίας δεδομένων και θα πρέπει οι εποπτικές αρχές να είναι έτοιμες να επιτελέσουν αυτό το έργο στον τομέα θέση σε ισχύ. Επίσης τώρα μας απασχολεί και το γενικότερο θέμα του κατεπήγοντος και καμία ρυθμιστική αρχή δεν ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχουν αυτοί οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί. Τώρα για το μέλλον για το 17 και μετά θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα και να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με ορισμένα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη που δεν τα κατανομάζω, δεν θέλω να τα ξεντροπιάσω, έχουν λιγότερο ε, ενδιαφέρον να θέσουν σε ισχύ ε, τη νέα νομοθεσία. Γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλη εργασία και σε αυτό το τομέα. Ε, σε σχέση με τη Γενική Συμφωνία ε, PNR και TTIP, καταρχήν να σταθώ στο TTIP γιατί υποβλήθηκαν αρκετές ερωτήσεις κατά πόσο δηλαδή η απόφαση επηρεάζει την ε, δική μας κρίση για το TTIP και την προστασία των δεδομένων, το PNR. Εγώ δεν θα είμαι ενεργό μέρος των διαπραγματεύσεων ε, για το TTIP διαφέρει από τις διαπραγματεύσεις ασφαλούς ε, λιμένα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι για την ε, μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Λάβουμε υπόψη δηλαδή και το σύστημα των ΙΠΑ, το νομικό σύστημα για τη Γενική Συμφωνία Umbrella Agreement, ε, εδώ είχαμε μία απόφαση επάρκειας που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αντίθετα, η Γενική Συμφωνία θέτει υψηλά, υψηλά τον πύχη για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια και της συνεργασίας της δικαιοσύνης ήπα Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν νομίζουμε ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις ε, της αποφάσεις της του δικαστηρίου. Σε σχέση με την Umbrella Agreement θα ήθελα να τονίσω και πάλι τις αποφάσεις για τη Γενική Συμφωνία μέσα στα πλαίσια και της συμφωνίας από το Κογκρέσο. Ο κύριος Σόλμπρεχτ υπέβαλε επίσης ένα ερώτημα. Ένα από τα θέματα ήταν οι υπηρεσίες πληροφοριών και η προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απασχολεί την απόφαση του δικαστηρίου. Όπως ξέρετε, εδώ μιλάμε για θέματα εθνικής ασφαλείας που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών ε, μελών. Και αυτό αφορά και τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει ε, για τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο. Και σε σχέση με ζητήματα δημόσιας τάξης ε, ασφάλειας και ούτω καθεξής, άρθρο 3 της οδηγίας 9546. Αλλά δεν πρόκειται για γενική εξαίρεση ιδιαίτερα ως προς την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η εθνική ασφάλεια ε, δεν μπορεί να γίνει επίκληση της εθνικής ασφάλειας παντού. Θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της αναλογικότητας, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις ε, παραμέτρους αναλογικότητας που ε, είναι αναγκαίες για θέματα συστήματος πληροφοριών και διάδοσης δεδομένων. Ο, ως προς το PNR και τις συμφωνίες TFTP υπάρχουν ε, δικλίδες ε, ασφαλείας σε σχέση με, την, ε, τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τις αρχές των ΙΠΑ. Και αυτό αφορά και τους Ευρωπαίους πολίτες που μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Αυτό το σχετίζεται με την προαπέτηση του δικαστηρίου έτσι ώστε η ε, μεταφορά δεδομένων να παρέχει εγγυήσεις για να μην παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και αυτό αφορά και τα, τις δημόσιες αρχές των ΗΠΑ. Δηλαδή όταν υπάρχει συλλογή δεδομένων για άλλους στόχους από αυτούς που είναι απολύτως αναγκαίοι επιπρόσθετα, όπως απαιτεί το δικαστήριο, και οι δύο διευθετήσεις αφορούν συνεχή εποπτεία του συστήματος και η αξιολόγηση της συμφωνίας ε, PNR θα γίνει του χρόνου. Το 2013 ε, αναθεωρήθηκε και το 13 και το 15 για το TFTP ε, θα γίνει η αναθεώρηση του χρόνου. Γιατί η προηγούμενη έγινε το 13. Νομίζω ότι ήδη μίλησα αυτό που προαναφέρατε εσείς. Προσπαθ, πούμε να ε, βελτιώσουμε τη συμφωνία του ασφαλούς ε, λιμένα. Ακόμα και πριν από την απόφαση του δικαστηρίου ε, μιλήσατε για ένα χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τα τέλη του Μαΐου ήταν η αρχική προθεσμία, αν το θυμόσαστε, αλλά δεν είχαμε όλα τα δεδομένα και έπρεπε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και το καλοκαίρι. Νομίζω ότι υπήρξε καλύτερη εποπτεία του, του πλαισίου από τις ΕΠΑ κατά την μεταφορά δεδομένων. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία πώς αντιμετωπίζονται οι καταναλωτές από τις μεγάλες επιχειρήσεις και επίσης υπάρχουν μηχανισμοί προσφυγής στη δικαιοσύνη χωρίς ε, δικαστικά έξοδα. Επίσης ε, το καθεστώς των μεταφορών, το θέμα της ευθύνης. και ο πλέον ενεργός ρόλος ε, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών προστασίας δεδομένων που υποβάλλουν τα αιτήματά τους στο Ομοσπονδιακό Εμπορικό Επιμελητήριο για τον ασφαλή λιμένα. Και μίλησα και για την ετήσια αναθεώρηση για την σωστή χρήση του ασφαλούς λιμένα γιατί θα πρέπει να έχουμε να κάνουμε με πολύ καθαρές διαδικασίες και ε, διασφαλίσεις και μηχανισμούς διασφάλισης. Τώρα, σε σχέση με την επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, ε, την, την ανακοίνωσή μας, με συγχωρείτε, για τις επιχειρήσεις, ε, αυτό θα είναι ένα ενδιάμεσο μέτρο, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και θα υπάρχουν και οι διατάξεις που έχουν προσυμφωνηθεί γιατί αυτό που έχει σημασία είναι οι αρχές προστασίας των δεδομένων που είναι οι αρχές θέσεις εφαρμογή να το κάνουν αυτό. Όμως ποια είναι η υποχρέωση της οδηγίας που έχει τεθεί σε ισχύ και ποιες είναι και οι εναλλακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Υπήρξε και μία ερώτηση για τις ΜΜΕ, για την προστασία τους. Ίσως ε, δεν αναφέρθηκα στην, ε, στις επίγραμ, στους επιγραμμικούς λόγους ε, μίσους, online δηλαδή. Αυτό είναι ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Ξέρετε ότι οργανώσαμε ένα ετήσιο συμπόσιο για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και είχαμε και τη διάσκεψη για τη ριζοσπαστικοποίηση ανθρώπων που μετά μεταβαίνουν στη Συρία, στη Μέση Ανατολή και επανέρχονται ως μαχητές, ως ξένοι μαχητές. Είδαμε με τα κράτη-μέλη ότι ένα 15% αυτών των νέων ε, ρίζοσπαστικοποιούνται στις φυλακές. Δυστυχώς οι φυλακές είναι μία από τις πηγές ριζοσπαστικοποίησης. Η πλειοψηφία όμως ακολουθεί αυτή τη διαδικασία online. Εκεί εκπαιδεύεται. Γι' αυτό προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πλήρως την συμφωνία πλαίσιο του 2008 που ε, τονίζει το γεγονός ότι οι λόγοι μίσους που μπορούν να οδηγήσουν σε ε, ρατσιστικά εγκλήματα με βάση τις θρησκευτικέ προτιμήσεις, ε, το χρώμα του δέρματος και ούτω καθεξής, όλοι αυτοί οι λόγοι θα πρέπει να διαγραφούν από τους ιστότοπους καθώς και ορισμένες εκφράσεις που μπορούν να επιταχύνουν τις τρομοκρατικές ε, βιοπραγίες. Αυτό εντάσσεται στο ποινικό δίκαιο και συμφωνήσαμε και με τους Υπουργούς ε, Δικαιοσύνης ότι θα πρέπει να κατανοούν τον κίνδυνο που ελοχεύει στην Ευρώπη σε σχέση και με την κρίση των προσφύγων και θα πρέπει να επιβάλλουμε τον νόμο. Όταν μιλάμε για την καταπολέμηση του ρατσισμού και τους, το λόγο μίσους, ε, δεν μιλώ για νέα νομοθεσία, μιλώ για την εφαρμογή του προϋπάρχοντος νόμου μέσα στα πλαίσια του ποινικού δικαίου. Ήδη συζήτησα με τους ε, διαδικτυακούς παρόχους κατανοούν ότι είναι μέρος του προβλήματος και θα πρέπει να είναι και μέρος της επίλυσης του προβλήματος. Κοινωνεί δηλαδή της λύσης του προβλήματος. Από ό,τι κατάλαβα κατανοούν τις νομικές τους υποχρεώσεις και έχουν πάρει πολύ σοβαρά και την κοινωνική τους ευθύνη, τον κοινωνικό τους ρόλο σε αυτή την εργασία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις συζητήσεις και με τους παρόχους και σε συνεργασία με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των μεγάλων αυτών απειλών. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να καλύψω όλα τα ζητήματα, ελπίζω να μην παρέλειψα κάτι. Εάν δεν λάβατε απάντηση, να μου το πείτε. Μπορούμε να ακολουθήσουμε και τη γραπτή διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Um, <clears throat> Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Δεν έχουμε χρόνο για πρόσθετες ερωτήσεις. Το χαρτοφυλάκιό σας ε, είναι πολύ ευρύ, πολύ πλούσιο. Ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας που κάνετε, ε, η δουλειά που κάνετε σε διάφορα άλλα θέματα κατά τη, με την αντίγραφη των διακρίσεων κλπ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά σας είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό το θέμα που συζητήσαμε σήμερα ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο να συνεχίσουμε, αλλά ε, οι, οι συνάδελφοι ρώτησαν τα εξής. Θέλετε να ξαναγυρίσετε, ε, ε σκοπεύετε να ξαναγυρίσετε στις 10 Δεκεμβρίου. Ε, συζητήσαμε την απόφαση για την προστασία των δεδομένων σήμερα. Είναι διαφορετική και από πλευράς περιεχομένου αλλά και από πλευράς ιστορικότητας. Ε, είναι μια πολύ σαφής απόφαση παρόλο που δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά ποιες θα είναι οι συνέπειες της. Οπότε θα πρέπει να την εφαρμόσουμε, να συμμορφωθούμε. Οπότε δεν θα ήταν λάθος να σας ζητήσουμε όταν ξανάρθετε το Δεκέμβρη να είστε σαφείς σε ό,τι αφορά την θέση της Κομισιόν. Σαφώς οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ηθική υποχρέωση να μετακινηθούν. Εμείς από την άλλη μεριά θα σας ζητήσουμε να μας ενημερώσετε για το τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Ένα. Δεύτερον, η Κομισιόν είναι θεματοφυλάκας των συνθήκων και πολλοί ρώτησαν, και ο Σκύρκο για παράδειγμα, ρώτησε τι, θα, τι μπορεί να πει και δεν μπορεί να πει το δικαστήριο. Όμως εσείς είστε ο θεματοφύλακας των συνθήκων. Οπότε όταν επιστρέψετε σε εμάς ε, θα μπορούσατε να ε, μας δώσετε μια ιδέα για το τι συνέπειες θα έχει αυτή η απόφαση ε, να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, το αν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για την ε, συμφωνία περί διαβίωσης χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων και λοιπά, ε, χωρίς να μπούμε σε ειδικέ συμφωνίες ενδεχομένω, αλλά μια πιο γενική αξιολόγηση. Το ζήτησαν και συνάλφοι, θέλουμε βεβαιότητα για τους πολίτες μας, θέλουμε βεβαιότητα, νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε σήμερα αλλά όταν επιστρέψετε στην Επιτροπή μας θα ήθελα αυτά να τα έχετε υπόψη για να μας ενημερώσετε. Ας έχουμε μια πολύ πιο ε, ε μεγάλη ασφάλεια, μια νομική βεβαιότητα και μια ε, μεγαλύτερη σαφήνεια στις απόψεις σας. Αυτά συναδελφοί, ας κλείσουμε. Θα συνεργαστούμε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, που δεν είναι ημερομηνία που απέχει και πολύ. Είναι και πολλή δουλειά έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε. Έτσι ώστε όλοι να κατανοήσουμε τις συνέπειες αυτής της απόφασης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και ευχαριστώ πολύ και για τις ερωτήσεις σας. Έχουμε και την συνάντηση των συντονιστών αμέσως μετά. Ευχαριστώ Επιτροπέ.